υπάρξουν και που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μελών ε, που ε, συνθέτουν το Κοινοβούλιο, δηλαδή 376. Σύμφωνα με το άρθρο 178, παράγραφος 3 του κανονισμού, για να διαπιστωθεί η επίτευξη των απαραίτητων δύο τρίτων υπολογίζονται μόνο οι ψήφοι οι οποίοι ε, ε, ε, είναι υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης προτάσεως. Υπάρχει μόνο υπέρ και κατά. θα συμπεριληφθούν στο πινακάκι που έχετε μπροστά σας και οι αποχές αλλά οι ψήφοι που θα ληφθούν η υπόψη είναι μόνο αυτές που συνοδεύονται από το συν και το πλην. Σύμφωνα με το άρθρο λοιπόν 180 παράγραφος 2 ε, προβλέπεται ε, να υπάρξει μυστική ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν, θα αρχίσουμε την ψηφοφορία. Κάποιος έχει στήσει το λόγο. Ο κύριος Λεγκούτκο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε ε, το άρθρο 184α για να διευκρινίσουμε την ψηφοφορία. Αψηφείτε τα δικαιώματα εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν αποχή. Ρωτήσαμε τις υπηρεσίες και είπατε ότι ε, οι αποχές δεν θα συμπεριληφθούν στην καταμέτρηση. Διαμαρτύρομαι εντόνως. Το άρθρο 21 ε, δεν είναι το ίδια η διαδικασία με την εκλογή των ε, αντιπροέδρων και η αποχή είναι εξίσου έγκυρη ψήφο όπω οποιαδήποτε άλλη ψήφο και είναι καθιερωμένη πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλουν υπόψη και οι αποχέ. Κύριε Πρόεδρε, επιμένω ε, από σεβασμό προ την κοινοβουλευτική δημοκρατία να λάβετε υπόψη και τι αποχέ στην καταμέτρηση έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων. Ο κύριος Σανέσκι δεν είχε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην Ολομέλεια, άκρος παράτυπο, και τώρα αφαιρείται και τις αποχές από την καταμέτρηση. Επίσης παράτυπο, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού, Ναι, η πρώτη φορά που γίνεται μια ψηφοφορία με βάση το άρθρο 21 και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ε, επικρατούσα γενική ε, ερμηνεία η οποία δίδεται σε όλες τις ψηφοφορίες γύρω από τα θέματα αυτά. Και για την εκλογή των προέδρων και των αντιπροέδρων δεν υπολογίζονται οι αποχές. Και σε σχέση με την έγκριση ουδήποτε κειμένου ή ασδήποτε προτάσεως, στα πλαίσια του υπολογισμού των ψήφων λαμβάνονται υπόψη μόνο ε, ε, τα υπέρ και τα κατά εκτός και εάν προτείνεται μια ειδική πλειοψηφία. Καμία συνθήκη όμως δεν προβλέπει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση και γι' αυτό εγώ διερμηνεύω ευραίως το 178 και όλους τους άλλους κανόνες οι οποίοι ανέκαθεν διακυβέρνησαν την εκλογή των προσώπων σε θέσεις στο Κοινοβούλιο. Θα ερμηνεύσω τον κανονισμό λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και επιβεβαιώνω ότι οι ψήφοι που θα ληφθούν υπόψη είναι οι υπέρ και η κατά και μόνον αυτή ο κύριος Κόρμπετ. Ήμουν εισηγητής για αυτόν τον κανόνα όταν εισήχθη στους, ε, στον εσωτερικό μας κανονισμό πριν από πολλά χρόνια και επιβεβαιώνω ότι η δική σας ερμηνεία είναι ακριβώς, αντιστοιχεί ακριβώς την πρόθεσή μας. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε τώρα. Μυστική ψηφοφορία. Θυμίζω ότι απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων μόνο υπέρ και κατά θα ληφθεί υπόψη. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Η πρόταση λοιπόν γίνεται δεκτή, λέει ο πρόεδρο. Θα περάσουμε τώρα στην έκθεση Ούμπνερ και Σίλβα Περέιρα για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Άρθρο 3, παράγραφος 1, ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. il voto è chiuso il testo è respinto απερίφθη τροπολογία 3 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απερίφθη αρχικό κείμενο ονομαστική κλίση ψηφίζεται τέλος Δεκτό. Τέσσερα Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. παράγραφος 4, άρθρο 1, τροπολογία 5, 18, 27, 39, ονομαστική κλίση, ψηφίζεται. Πέραση στις Δεκτό. Άρθρο 5, Αρχικό κείμενο ψηφίζεται ονομαστική κρίση. Πέρα στις Δεκτό. Στο 3, 16D και 26D ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Περνάμε στην πρόταση αποφάσεως. Ποιοι είναι υπέρ. Δεν είναι ονομαστική κλίση. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ της ε, προτάσεως αποφάσεως. Κατά. Αποχές δεκτή. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο βεβαίως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος. Μπρέσο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δημιουργήσατε μια κάποια σύγχυση. Δεν εξηγήσατε τι συμβαίνει. Δεν ήξερε ο κόσμος τι ακριβώς ψήφιζε. Είναι σαφές αυτό. Εμείς έχουμε μπροστά μας κατάλογο ψηφοφοριών και εσείς δεν εξηγήσατε το τι ψηφίζαμε. Κυρία Μπρέσο, Παρακαλώ, αν με ακούσετε ε, θα απαντήσω. Όχι, λέει η κυρία Μπέσου. Ευχαριστώ. Δεν εξηγήσατε, δεν είπατε ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το 4 καταπίπτουν. Δεν το είπατε αυτό ότι έχουν καταπέσει. Εμείς νομίσαμε ότι ψηφίζαμε αυτό και όχι το άρθρο 5. Δεν το είπατε, δεν το εξηγήσατε, δεν το καταλάβαμε. Κοιτάξτε στον κατάλογο που έχετε μπροστά σας λέγεται ότι στην περίπτωση που γίνουν δεκτές οι τροπολογίες αυτές καταπίπτουν οι 2 και τρία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Μίλησα για συγκεκριμένες προτάσεις. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Μπρέσο. Ομιλώ την Ιταλική, είναι η δική σας μητρική γλώσσα, πρέπει να με κατανοείτε περισσότερο από τους υπόλοιπους τουλάχιστον. Κάβα. Κοιτάξτε πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε μπλέξει εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε για μία ακόμη φορά την πρόταση αποφάσεως. Έχει ήδη ελεγχθεί αυτό και έχει ολοκληρωθεί. Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 5 το οποίο τέθηκε σε ψηφοφορία αμέσως μετά την υιοθέτηση του 4.1 ψηφίστηκε από πολλούς από μας κατά της του καταλόγου γιατί δεν γνωρίζαμε ότι επρόκειται για το άρθρο 5 και έτσι κι αλλιώς και ο πίνακας έλεγε άλλα πράγματα εμείς ζητάμε μία απλή επανάληψη της ψηφοφορίας του άρθρου 5 και να συνεχίσουμε αμέσως με τα κανονικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα θα βοηθήσει πολλούς συναδέλφους να ψηφίσουν με τον σωστό τρόπο. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί χτυπάτε το τραπέζι και γιατί χειροκροτείτε. Εγώ ήμουν σαφής σχετικά με την συγκεκριμένη τροπολογία. Ο πίνακας έλεγε τέσσερα, όχι πέντε. ο capito, ο capito. Κατάλαβα λοιπόν, μου είπαν εδώ, εγώ δεν βλέπω τον πίνακα, ότι μπορεί να έχει υπάρξει λάθος στον πίνακα σχετικά με το άρθρο 4 και το άρθρο 5. Θα ψηφίσουμε εκ νέου λοιπόν το άρθρο 5. Το αρχικό κείμενο του άρθρου 5. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. με να πίνω νερό. Πέρα τη ψηφοφορία έγινε δεκτό το κείμενο. Περνάμε τώρα λοιπόν 16D και 26D ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. Καταπίπτει η τροπολογία υπαριθμών 38. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση αποφάσεως. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος. Η ηλεκτρονικός έλεγχος για την προηγούμενη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. Πρόταση ψηφίσματος. Παράγραφος 1. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Αρχικό κείμενο στην παράγραφο 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Παράγραφος 5. Το αρχικό σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τροπολογία 15 σε δύο τμήματα. Α, όχι, έχει καταπέσει και η 15. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 41. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 ψηφίζεται. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, λέει ο Πρόεδρος. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 2. Στην 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23 και 36. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτό. Καταπίπτει το αρχικό κείμενο. Περνάμε τώρα στην 7. Μετά την παράγραφο 9 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 24 και 42 στην 13. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 14-25 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Μετά την παράγραφο 15 έχουμε την 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 6. Πέρα τη ψηφοφορία. Απερίφθη. Λοιπόν, πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά του ΣΥ. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μετά το ΣΥ έχουμε το 8. και είναι υπέρ. Ψηφίζεται μάλλον. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη στο F αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το πρώτο ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Μετά το F έχουμε το 9 ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Το 10 και το 11 καταπίπτουν, οπότε περνάμε στο G, 19D, ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Καταπίπτει το 30. Το 31 λοιπόν ονομαστική κλίση ψηφίζεται στο H. Τέλος. Απερίφθη. 32 ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Μετά το H έχουμε το 12 ονομαστική κλίση. Άρχεται. Τέλος. Απερίφθη. 20 στο I. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτό. Μετά το I έχω την 13. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απέχουν Απερίφθη. Λοιπόν, 21 αντί και 34 αντί ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην 14D Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική κλίση ψηφίζεται. 18 συγχαρητήρια στους συνεισηγητές. Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκονσάλες Πόνς για την αναθεώρηση της Συμφωνίας Πλαισίου. Παράγραφος 1, τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 18 ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Παράγραφος 2. Αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 3. Η τροπολογία 3. Κλίση ονομαστική ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη 4D άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 5. Ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτό. Επτά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται. πέρα στις ψηφοφορίες το κείμενο γίνεται δεκτό. Περνάμε τώρα στην 7 ε, ονομαστική κλίση. Ψηφίζεται. Πέραση τη ψηφοφορίες. Απερίφθη. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές απερίφθη. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 9, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 11. Ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απερίφθη. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτό δεύτερο τμήμα, ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτό. Μετά την 11 έχω την τροπολογία 12, ονομαστική κλίση, ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Στην 12 έχω την 16, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε τώρα στην 10 και είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Τροπολογία 1 για μια στιγμή. Μεσολαβή 13. Λοιπόν, ονομαστική κλίση ψηφίζεται για την 13. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ένα τροπολογία ονομαστική κλίση ψηφίζεται. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν δεκτό. Το F αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 15 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 17 ονομαστική κλίση Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Αρχικό κείμενο στο J. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το αρχικό κείμενο. Πέρας ψηφοφορίας. Το κείμενο γίνεται δεκτό. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 συγχαρητήρια στον κύριο Κονσάλες Πόνς. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Κοράο, ονομαστική κλίση, ενία ψηφοφορία, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακολουθεί τώρα η πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των μειονοτήτων και απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία και μοναδική ψηφοφορία, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Προχωρούμε. Προσθήκη τη Σρι Λάγκα, του Τρινιδάδ και τον Πάγκο και τη Τινησία στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου Κυρία Επίτροπε, ε, κυρία Γιούροβα, επιθυμείτε να λάβετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, όλοι αναγνωρίζουμε τις κοινέ ευθύνε στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εργαστεί ιδιαίτερα σκληρά για να βελτιωθεί η οδηγία ένα, κατά του ξεπλήματος ε, χρήματος και να βελτιωθεί και το νομικό πλαίσιο. Ε, η, η πράξη που θα ψηφίσετε αφορά την, ε, την Ισία, η οποία είναι αναγνωρισμένη στενή σύμμαχος και συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η πράξη δεν θα υποσκάψει οποιαδήποτε πολιτική ή χρηματική οικονομική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την Τινησία. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο της Τινησίας τις τελευταίες εβδομάδες. Η Κομισιόν θα στηρίξει στενά την τινησια αναγνωριζουμε την προοδο της τινησιας στις τελευταιες εβδομαδες προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα δράσης που έχει συμφωνηθεί και θα στηρίξει την, ε, task force, ε, την οικονομική task force ε, το Δεκέμβρη. Θα είμαστε σε στενή επαφή με τους τινήσιους φίλους σε ό,τι, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Θα δώσουμε βοήθεια στην Τινησία έτσι ώστε να ε, απαλληφθούν οι, υπάρχουσες, ελάχιστες υπάρχουσες αδυναμίες. η απομάκρυση από την λίστα ελπίζουμε θα γίνει από την ΦΑΤΦ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα σύντομα. Είμαι πεπισμένη ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας η Τινησία θα αποτελέσει υπόδειγμα για άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες και τη δέσμευση προσήλωσή τους. Τέλος, να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν εργάζεται ε, επί μια συστημικής λύσης έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τη δική της ανεξάρτητη ανάλυση ό,τι αφορά τον κίνδυνο που αποτελούν τρίτες χώρες για να προστατεύσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θυμίζω ότι ποιος θέλει, κύριε Βερζιά. Κύριε Βερζιά, παρακαλώ διαδικαστικό είναι, παρακαλώ, βάσει ποιο άρθρο του κανονισμού. Κυρία Πρόεδρε, εγώ έχω συντάξει την αντίρρηση και έλαβε το λόγο η κυρία Επίτροπο. Θα ήθελα μόνο να πω στου συναδέλφου ότι η κυρία Επίτροπο δεν προσέθεσε τίποτα στα όσα μα είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ και τη Δευτέρα στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να προσθέσω σας παρακαλώ. Τώρα δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση, ούτε να την επαναλάβουμε, λέει η Πρόεδρος. Έχει λάβει χώρα. Λοιπόν, ψηφίζουμε παρακαλώ, λέει η κυρία Γκέπχαρτ. Και θυμίζω ότι απαιτείται πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου για να εγκριθεί. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Νομίζω ότι δεν έχει εγκριθεί αντίρρηση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα το επαληθεύσουμε απολύτω. Φυσικά, παρακαλώ, αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασα. 357 υπέρ απορρίπτεται διότι η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών είναι 376. Προχωρούμε. Πρόταση ψηφίσματος μηδενική ανοχή στο θέμα του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ. Παράγραφος 4. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ψήφι Το αρχικό κειμένου. Κατά εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί παράγραφος 13, τροπολογία 3, με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα προχωρούμε στην ψήφιση του αρχικού κειμένου. Είναι και αυτή η ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα για την παράγραφο 13. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 4. Ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολόγια παριθμών 5. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολόγια υπαρθών 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολόγια παριθμένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία πε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο τώρα σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τελειώσαν οι ψηφοφορίες εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε με ταχύτερο ρυθμό και λιγότερο θόρυβο. Θα πω και ονόματα τώρα, κύριε Ελίζα και κυρία Γκυγιόμ.